όργανο που δεν εξασφαλίζει δίκαιη κατανομή, που θα αυξήσει τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ε, κλάδου και θα μπορεί να, να χρηματοδοτεί ακόμη και την αμυντική βιομηχανία, κάτι που είναι πραγματικά πολύ λυπηρό. Ο κύριος Ιγνάσιο Φαρία έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον κύριο Ζουζέ Μανουέλ Φερνάντες για το έργο του στο InvestEU. Ε, Στόχο είναι να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη και να απλουστευτεί αυτό το όργανο με το συνδυασμό των ε, ε, επιμέρους χρηματοδοτικών μέσων. Επίσης, μια εποχή που μας λείπουν οι ψηλέ επενδύσει για, για το καλύτερο μέλλον της Ευρώπης. Θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την υποστήριξη του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Σίγουρα με το InvestEU θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε τις βασικές στρατηγικές ε, και να αξιοποιήσουμε τη συμπληρωματικότητα με τα άλλα χρηματοδοτικά μέσα και των κρατών μελών. Έτσι, μικρές χώρες όπως η Πορτογαλία θα έχουν πρόσβαση σε περισσότερα προγράμματα ε, και που μέχρι στιγμής δεν ε, συγκέντρωσαν επενδύσεις ή ενδιαφέρον ιδιωτικού κλάδου. Ελπίζω να βρεθούν τα κατάλληλα προγράμματα για να περιορίσουμε τις κλιματικές αλλαγές και την αστάθεια της οικονομίας και να προωθήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βιοπικιλότητα. Ευχαριστώ. Η κυρία Βυσνιεύσκα έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, το πρόγραμμα InvestEU μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την τόνωση των επενδύσεων στις περιοχές που θα περάσουν έναν ενεργειακό μετασχηματισμό. Στη γνωμοδότηση της ΕΒΗ αναφέρουμε ότι οι επενδύσεις του InvestEU θα πρέπει ε, να ε, δοθούν ιδιαίτερα σε περιφέρειες που προβαίνουν σε ένα μετασχηματισμό που σχετίζεται με τις περιβαλλοντικές αλλαγές ε, και κυρίως την αλλαγή των υποδομών τους. Η πρώτη ευρωπαϊκή Επιτροπής δεν περιλαμβάνει ρητά αυτό το στόχο. Ερωτώ λοιπόν, από το πρόγραμμα InvestEU θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε και επενδύσεις ε, σε, παραγωγές, ε, σε περιοχές ε, που ήταν ε, κατά παράδοση ανθρακοπαραγωγές περιοχέ τη Ένωση, ώστε να πραγματοποιήσουν αυτό τον ενεργειακό μετασχηματισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ευρωπαϊκή πολιτική. Γιατί χώρε που έχουν ε, ενεργειακό μείγμα που στηρίζεται στον άνθρακα θα ε, πρέπει να καταβάλουν τεράστιο κόστο για να προσαρμοστούν στα περιβαλλοντικά κριτήρια. Καλό ήταν λοιπόν αυτέ οι χώρε να μπορέσουν να αποφεληθούν από τα κονδύλια του InvestEU. Και το λέω αυτό Πολωνέζα, γιατί ενδιαφέρει ιδιαίτερα την πατρίδα μου η πρόσβαση σε τέτοιε επενδύσει. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μάλη, είναι τελευταία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του συνηγητέ, Φερνάντε και Γουαλτιέρη ε, και να χαιρετήσω ιδιαίτερος ε, τον Αντιπρόεδρο Κατάινεν που έκανε περιοδία σε όλες τις ε, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Ελπίζω την επιτυχία του ΕΦΣΙ να την μεταλαμπαδεύσουμε και στο νέο πρόγραμμα του InvestEU. Εγώ όταν ασχολήθηκα με το πρόγραμμα στρατηγικών επενδύσεων διαπίστωσα πόσο σημαντική είναι η προεργασία, η προετοιμασία των προγραμμάτων ε, πώς θα πρέπει να ετοιμάσουμε τα κράτη-μέλη για να υποβάλουν αξιόλογα προγράμματα. Και αυτό θα πρέπει να κάνουμε και στο InvestEU. Να δώσουμε βοήθεια τεχνική και κυρίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες που δεν έχουν τις απαραίτητες διοικητικές ικανότητες να προετοιμάζουν τα προγράμματα και να συμμετέχουν και να υποφελούνται από αυτό το πρόγραμμα. Αυτό είναι μια σημαντική προϋπόθεση. Δεύτερο σημαντικό θέμα είναι να ε, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους, όχι μόνο τους οικονομικούς, αλλά να χρηματοδοτούμε καινοτόμε επιχειρήσεις, ε, ε, καινοτομία, startups, για να συμβάλλουν σε μια πιο βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ και τώρα το λόγο έχει εκ νέου ο κύριος Κατάινεν και εν συνεχεία οι δύο συγγητές παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενθαρρυντικά τα λόγια που ακούστηκαν στη συζήτηση να απαντήσω σε κάποιες ανησυχίες, ερωτήσεις και σχόλια και ιδέες που ακούστηκαν από τα αξιότιμα μέλη. Πρώτα απ' όλα, το Ταμείο InvestEU καθοδηγείται περισσότερο τις πολιτικές εν συγκρίση με το ΕΦΣΙ περισσότερο από ότι το ΕΦΣΙ. Δεν σημαίνει ότι γίνεται πολιτική επιλογή των προγραμμάτων και των έργων. Επιλέγονται βάσει της ποιότητας ε, των σχεδίων και εξετάζεται κατά πόσο το ΕΦΣΙ μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία. Η ιδέα είναι να καλύπτονται πολιτικές, όπως η αλλαγή του κλίματος, η βελτίωση της ψηφιοποίησης, η αύξηση της χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης σε κάποια κράτη-μέλη. Αυτό εννοώ όταν λέω ότι καθοδηγείται περισσότερο από πολιτικές. Δεύτερον, βασική ιδέα του ΕΦΣΥ θα παραμείνει. Το InvestEU ε, είναι εθελοντικό, κανείς δεν υποχρεώνεται να χρησιμοποιήσει το ΕΦΣΥ αν δεν θέλει να το χρησιμοποιήσει. Και αντίστροφα. Μπορεί να έχει σηματοδότηση εύση αν κάνει την αίτηση. Τρίτο στοιχείο. Η ιδέα του ΕΦΣΙ είναι να χρησιμοποιεί ιδιωτικούς πόρους για επενδύσεις από τα ταπεζικούς λογαριασμούς για επενδύσεις που δημιουργεί ανταγωνιστικότητα θέση απασχόλησης και επιτυχαίνει τους στόχους πολιτικής ομαδοποιώντας 13 εφιστάμενα χρηματοστικά μέσα συναθίζοντας τα αυτά ο τελικός χρήστης είναι πιο, εύχριστο, είναι, είναι πιο εύκολα χρησιμοποιήσει το InvestEU. Δεν χρειάζεται να γνωρίζει κανεί 13 διαφορετικούς ε, τρόπου και διαδικασίε και πόρου ο κάθε χρήστη. Ο Χρήστη πρέπει να ξέρει ότι υπάρχει το ταμείο InvestEU που μπορεί να δώσει πόρους και να χρηματοδοτήσει ποικιλοτρόπω τα προγράμματά σου. Πέρα από αυτό το συνδυασμό και από τη συνάθρηση 13 ταμείων θα έχουμε και 13 διαφορετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Για τον τελικό χρήστη, η, το να ζητήσει τεχνική αρρωγή είναι πολύ πιο εύκολο. Μέσω του InvestEU θα δώσουμε 25% των εγγύσεων ανάλογα με τη ζήτηση από άλλους από άλλα χρηματοσυντικά ιδρύματα εκτό τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι πολύτιμο εταίρο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο μέλλον. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε όμω και καινοτομίε χρηματοσυντικέ τομέ. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν πάντα σε θέση ή δεν επιθυμεί να επενδύσει και να καλύψει όλα τα έργα. Οι διάφορες εθνικές τράπεζε προώθηση, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να το κάνει. Αυτή, αυτό το ποσοστό το 25% ε, που έχει τεθεί θα δώσει προστιθέμενη αξία όσον αφορά τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Να επενθυμίσω κάτι στα αξιότιμα μέλη. Αν ενδιαφέρεστε και θέλετε να δείτε τα επιτέγματα του ΕΦΣΥ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΕΦΣΥ Μέσω του Google το βρίσκεται εύκολο. Ή πάτε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, φαίνεται κάθε πρόγραμμα που έχει εγκριθεί. Βάζετε τη χώρα σας και βλέπετε κατάλογο έργων που ήδη έχουν υπογραφεί στη χώρα σας. Το ΕΦΣΙ δεν ήταν επανάκια. Ούτε το Invest EU είναι το φάρμακο που γιατρεύει όλα τα πιθανά προβλήματα στον κόσμο. Είναι όμως πολύτιμο πρόσθετο εργαλείο επενδυτικό που μπορεί να εξυγχρονίσει την οικονομία μας, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να κάνει την οικονομία σφιβιώσιμη και να δώσει προστιθέμενη αξία και να συμβάλλει στην ευημερία των κοινωνιών μας. Τελευταίο σημείο για το ΕΦΣΥ. Κάτι που με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο, βλέποντας τα επιτεύγματα του ΕΦΣΥ, είναι να δω τι έγινε στις χώρες που ωφελήθηκαν περισσότερο από το ΕΦΣΙ. Αν δείτε τις επενδύσεις στο ΕΦΣΙ κατά ε, χώρα και ΑΕΠ αναχώρα, υπαριθμών ένα χρήστη είναι η Ελλάδα. Δεύτερον, δεύτερη είναι η Εστονία, τρίτη είναι η Πορτογαλία, τέταρτη η Ισπανία, πέμπτη η Λιθουανία, η Λετωνία είναι έκτη, η Βουλγαρία έβδομη, η Φιλανδία όγδοη, η Πολωνία ένατη και η Ιταλία δέκατη η χρηματοδότηση πήγε προς τη σωστή κατεύθυνση στους επιτοπλίστων, προς τις χώρες και περιοχές των χωρών αυτών που αντιμετώπισαν κάποιους οικονομικούς περιορισμούς και βλέποντας και την ποιότητα των έργων και των προγραμμάτων είναι εντυπωσιακά τα πράγματα. Έχουμε βελτίωση από όταν άρχισε το ΕΦΣΥ και είμαι σίγουρο ότι το InvestEU το ίδιο θα πετύχει στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στου αγορητέ, ο κ. Φερνάντε και μετά ο κ. Γκουαλτιέρη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ του συναδέλφου που έλαβαν μέρο στη συζήτηση. Ε, με εντυπωσιάζει που κάποιοι στράφηκαν κατά των ιδιωτικών επενδύσεων. Λίγοι ήταν βέβαια, αλλά παρόλα αυτά και αυτά τα ακούσαμε στην Ολομέλεια. Ε, Πολλέ επιχειρήσει όμω και μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι ιδιωτικέ. Και αυτό το πρόγραμμα, το InvestEU, δύναται και οφείλει να χρησιμοποιείται από τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές και έχει μεγαλύτερη προσθεθέμενη αξία. Είναι ένα επιπλέον χρηματοδοτικό εργαλείο για, την, ε, για τις επενδύσεις, ιδιαίτερα εκεί που υπάρχουν κενά στην αγορά εκεί που λείπουν οι επενδύσεις. Και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι κατανόητο. Αυτοί που από τη μια θέλουν ε, περισσότερες θέσεις απασχόλησης στρέφονται κατά κάποιων ε, μηχανισμών που τονώνει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Επίσης, ε, το InvestEU έχει έναν άξονα που ενισχύσαμε εμείς, που είναι ο άξονας των κοινωνικών, του κοινωνικών υπηρεσιών και υπάρχει και μια ειδική θηρίδα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Επίσης, α μην υπάρχει σύγχυση ε, για το τι προβλέπεται για τα κράτη-μέλη. Πέραν των 700 δισεκατομμύριων που προτείνουμε για τις επενδύσεις, με τις εγγύήσει περίπου 40 δισεκατομμύρια, υπάρχει δυνατότητα των κρατών μελών να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα InvestEU και να δώσουν εγγύηση ε, από τα διαρθρωτικά ταμεία, χωρίς μεταφορές, ε, γιατί α, υπάρχει ένα ποσοστό του Διευθυντικού Ταμείου που ανήκει στα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη μπορούν με το τριπλό α να αξιοποιήσουν την ευκαιρία αυτή και να αποφύγουν τις δυσκολίες που έχουν στα οικονομικά τους για να προβλέψουν επιπλέον επενδύσεις για συγκεκριμένα σχέδια. Φυσικά, σε ό,τι αφορά τη χρήση αυτής της θηρίδας, ε, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να χρηματοδοτήσουν τα σχέδια που θεωρούν τα πιο σημαντικά. Και ε, η ψηφοφορία στην Επιτροπή Προπολογισμών ήταν ε, συντριπτικά υπέρ των υπερμάχων της ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και υπέρ της στήρισης των υποσχέσεων που δώσαμε για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Φερνάντος, ο κύριο Γκουαλτιέρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ήταν πλούσια η συζήτηση και αντικατοπτρή συζήτηση την πολύ μεγάλη συνένεση του Κοινοβουλίου όσον αφορά το κείμενο το οποίο ενεκρίθη στις δύο επιτροπές, την ΕΚΟΝ και την Budget. Πιστεύω ότι ως διεφάνει και από την παρέμβαση του Αντιπροέδρου Κατάινεν, Έχουμε μπροστά μας μια θετική διαδικασία αυξητική. Το ΕΦΣΙ πετέλεσε μια επιτυχία, αλλά σίγουρα δεν μπόρεσε να χρησιμοποιήσει όλη τη δυναμικότητά του όσον αφορά την ποιότητα των επενδύσεων και τη δυνατότητα να καλύψει εις βάθος τις ελλείψεις της αγοράς. Το InvestEU, όπως προτείνεται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και όπως ευελτιώθη μάλιστα από το Ευρωκοινοβουλίο πιστεύω ότι καθορίζει σωστή ισορροπία μεταξύ ευελιξίας, προσανατολισμού βάση πολιτικής, λεπτομέρειας και ταυτόχρονα οικονομία κλίμακας επιτυγχάνει. Θεμελιώδης είναι η βεβαιότητα για τους πόρους και γι' αυτό ευχόμεθα και ελπίζουμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο να είναι στο ύψος των περιστάσεων, να μπορεί ποσοτικά να ενισχύσει την προσπάθεια πέρα από την ποιοτική αύξηση που πετυχαίνουμε στο κείμενο για το InvestEU. Η ομάδα μας θα ευθυγραμμιστεί απόλυτα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Επιτροπές και ελπίζω κάποιες τροπολογίες ε, επιβλαβής να μην ε, εγκριθούν για να δώσουμε ισχυρό μήνυμα όσον αφορά το πώ θέλουμε να πετύχουμε ε, την βιωσιμότητα ε, όσον αφορά την όλη προσπάθεια από πλευρά Κοινοβουλίου. Σα ευχαριστώ. Η πρόεδρο, ευχαριστούμε. Εδώ ολοκληρώθηκε η συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Και τώρα. Θέλω να καλωσορίσω θέρμα την Επίτροπο Μάλστρομ και να αποχαιρετήσω τον ε, Επίτροπο Κατάινεν. Ευχαριστώ όσου ε, συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση και περνάμε στην κοινή συζήτηση για την εφαρμογή των συμφωνιών εμπορίου ή σύνδεση στη Λατινική Αμερική. Μιλάμε για την Κολομβία και το Περού. Εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Κολομβίας και Περού. Η ε, είναι ο Σαντιάγο Φίσας αυτή είναι η πρώτη έκθεση και η δεύτερη έκθεση είναι έκθεση εφαρμογή σχετικά με τον εμπορικό πυλώνα τη συμφωνία Σύνδεση με την Κεντρική Αμερική με εισηγητή τον κύριο Μπέγκε. Καταρχάς λοιπόν έχουν το λόγο οι εισηγητέ Φίσα και Μπέγκε. Καταρχάς ο κύριος Φίσα τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώ ήρθατε, κυρία Επίτροπε. Η εμπορική συμφωνία που υπογράφηκε το 2013 μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση, Κολομβία και Περού εφαρμόστηκε προσωρινά την τελευταία πενταετία και μετά την αξιολόγηση ε, τη εφαρμογή και των σχέσεων των τριών χωρών, διαπιστώνουμε ότι ήταν μια υποφελή για όλου συμφωνία. Η εμπορική αυτή συμφωνία ξεπερνά ε, τις αμυγός εμπορικές πτυχές, γιατί προϋποθέτει μια σχέση που εδράζεται σε κοινέ αρχές και αξίες και σε διεθνή πρότυπα ε, κάτι που συνέβαλε πολύ θετικά στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη των συμβαλωμένων μερών. Επίση, πρόκειται για ένα εργαλείο που μα επιτρέπει να εμπεδώσουμε, να εδραιώσουμε μάλλον τη στρατηγική μα σχέση με τη Λατινική Αμερική, κάτι που είναι ζωτική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εμπορική αυτή συμφωνία συνέβαλε στην οικονομική σταθερότητα, τον εξυγχρονισμό και την ε, διαφοροποίηση των εξαγωγών ε, τη Κολομβία και του Πέρου προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό για τι δεύτερε χώρε να έχουν μια αγορά αναφορά πέραν των χωρών τη Λατινική Αμερική για να ε, έχουν διαφορετικού προορισμού για τι εξαγωγέ του. Χάρη στη συμφωνία αυτή, η Κολομβία και το Περού εξυγχρόνησαν και διαφοροποίησαν τι εξαγωγέ του ε, με θετικό αντίκτυπο για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει του. Αλλά θετικό ήταν ο αντίκτυπος και για τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει, γιατί βελτιώθηκε η πρόσβασή του στι αγορέ του Περού και Κολομβίας, όχι μόνο μέσω τη κατάργηση των δασμολογικών ε, των δασμών, αλλά και τη, λόγω της άρσης των μη δασμολογικών εμποδίων. Και γι' αυτό ε, καλό θα ήταν οι μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν το έπακρο το δυναμικό τέτοιου είδους εμπορικών συμφωνιών. Επίσης θετικά αξιολογούμε το γεγονός ότι προχωρήσαμε στην αναζήτηση λύσεων ε, για τους ε, υπάρχοντες εμπορικούς φραγμούς, ιδιαίτερα για τα ε, υγειονομικά και φυτογειονομικά θέματα. Βέβαια, το Περού και η Κολομβία θα πρέπει να λύσουν θέματα όπως πιστοποίηση κάποιων ε, γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατο, ε, θέμα γεωγραφικών ενδείξεων τη ευρωπαϊκή Ένωση. η φορολογια που εφαρμόζεται στα ενοπνευματόδη. Ε, χάρη στην συμφωνία αυτή προωθήσαμε κάποιου μηχανισμού συνεργασία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των κυβερνήσεων Κολομβία και Περού, ιδιαίτερα για εμπορικά θέματα και ζητήματα βιώσιμη ανάπτυξη. Στόχο μα θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση ε, των παγκόσμιων ε, διατάξεων για το περιβάλλον και τις εργασιακές συνθήκες. Και επειδή συνοδεύεται από δικό χάρτη, η Εμπορική Συμφωνία χρησιμεύσε για την παρακολούθηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων και μάλιστα διαπιστώνουμε πρόοδο στα θέματα αυτά από τις δύο χώρες, το Περού και την Κολομβία. Βέβαια, ακόμη υπάρχει δρόμος μπροστά μας. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ελευθερία ε, τους συνεταιρίζεστε, το δικαίωμα στις συλλογικές ε, διαπραγματεύσεις, ε, εργασιακές επιθεωρήσεις, καταπολέμηση της παιδικής εργασίας, της άτυπης εργασίας ή πρόθεση των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυβέρνηση τη Κολομβίας για την κατάπαυση του πυρός και την πάυση των εχθροπραξιών και τη συμφωνία με, τη, με τον Τάρκτικο των ΦΑΡΚ και επίση τη συμφωνία του ΟΣΑ τη 30 η Μαΐου που αναγνωρίζει τι σημαντικέ μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην Κολομβία. Επίση, θα ήθελα να εθαρρύνω το Περού να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις του στα πλαίσια του προγράμματος που έχει στον ΟΣΑ. Επίσης, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ε, τέτοια συμφωνία θα έπρεπε να είχαμε συνάψει με όλε τι χώρε του Συμφώνου των Άνδρων και με τη Βολιβία και τον Ισημερινό, που για πολιτικού λόγου ε, απέρριψαν τι διαπραγματεύσει. Χαίρομαι πάντω ε, που η σημερινό ζήτησε να προσχωρήσει το 2015, λαμβάνοντα υπόψη ποια θα ήταν τα πλεονεκτήματα για την οικονομία του. Και μάλιστα το Κοινοβούλιο του Ισημερινού το Δεκέμβριο του 2017 ενέκρινε την προσχώρηση του Ισημερινού. Θα πρέπει οι φίλες αυτές χώρες ε, να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους ε, και να συνεχίσουν την πρόοδό τους. Πάντως θα ήθελαμε να τους συγχαρούμε για τη μέχρι τώρα πρόοδο που έγινε και με την υποστήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μπέγκε έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η εκθέση αυτή για την εφαρμογή του εμπορικού πυλώνα Συμφωνία Σύνδεση με την Κεντρική Αμερική έγινε δεκτή στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου με μεγάλη πλειοψηφία. Σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, ε, το παγκόσμιο εμπόριο που θα βασίζεται σε κανόνες είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να φέρει περισσότερη σταθερότητα ε, στον κόσμο που αλλάζει. Στην έκθεση αυτή υπάρχουν και θετικά αλλά και ε, σχόλια τα οποία ε, δείχνουν κάποιες, ε, κάποιο προβληματισμό σε ό,τι αφορά αυτή τη συμφωνία σύνδεσης. Τρεις είναι οι πυλώνες. Δυστυχώς μέχρι σήμερα ε, παρότι τα κράτη της Κεντρική Αμερική έχουν από το 2013 υπερψηφίσει και επικυρώσει την ένεση. Δυστυχώ έχουμε τρία κράτα οποία ε, δεν έχουν ακόμη ε, επικυρώσει τα δύο από τα τρία σκέλη. Ε, και αυτό υπονομεύει και την αξιοπιστία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. σε ό,τι αφορά τους εταίρους μας από άλλες υπήρους, με τους θέλουμε να έχουμε συμφωνίες σύνδεσης ή άλλε εμπορικές συμφωνίες. Επομένως, ε, πρώτα απ' όλα, απευθύνω έκκληση στα τρία αυτά κράτη-μέλη να προχωρήσουν τάχιστα στην κύρωση αυτής της συμφωνίας ώστε να υπάρξει μια ισορροπημένη σχέση του εμπορικού πυλώνα, ε, του πυλώνα της συνεργασίας ε, και του πυλώνα του πολιτικού διαλόγου. Θέλω επίσης να πω πως η συμφωνία αυτή είναι η πρώτη συμφωνία μεταξύ περιφερειών αν θέλετε, με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής αυτές, ε, πρέπει να πω ότι βλέπουμε ότι έχουν διαφορετικές προκλήσεις και ιδιαιτερότητες ε, και μπορώ να σας αναφέρω ορισμένα πράγματα. Υπάρχουν κράτη όπου ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ενώ υπάρχουν άλλα κράτη που προχωρούν με πιο βραδείς ρυθμούς. Ταυτόχρονα βλέπουμε πως ε, υπάρχει και κάποια σύνδεση ε, με τις αλλαγές που γίνονται. Παραδείγματο χάρη στις χώρες όπως η Κωνσταντίνα που αυξήθηκε πολύ ο όγκος συναλλαγών, μετά είναι η Κωνσταντίνα και ο Παναμά. Από την άλλη ε, πλευρά βλέπουμε στην νοτιοανατολική Ασία να μειώνονται δραματικά οι εμπορικές συναλλαγές. Και είναι αυτά θέματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε. Βλέπουμε επίσης και σε, όπως και σε άλλες ε, εμπορικές συμφωνίες ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι άλλοι ε, εταίροι σε ό,τι αφορά τις, ε, τους δασμούς και τις άλλες ποσοστώσεις τις αξιοποιούν. ένα ένας τομέας που εστιάζουμε πολύ, ο πρωτογενής τομέας. Εκεί υπάρχουν πολλές εξαγωγές και νομίζω ότι εκεί πρέπει να σημειωθεί ακόμα μεγαλύτερη πρόοδος. Θα πρέπει να πω επίσης ότι υπάρχουν διάφοροι τομείς για τους οποίους πρέπει να γίνει πολύ πιο εντατική συζήτηση, όπως είναι η παροχή υπηρεσιών. Η Επίτροπος Μάλστρομ χρειάζεται να αναλάβει δράση. Από αυτού απευθύνω έκκληση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κεντροαμερικανικά κράτη να εφαρμόσουν πλήρως και να κυρώσουν και την ε, Διεθνή Περιβαλλοντική Συμφωνία του Παρισιού και να τηρήσουν τις σχετικές δεσμεύσεις. Επαναλαμβάνω ότι πρέπει να εφαρμοστούν και οι διατάξεις ε, των συμφωνιών ε, και συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας εκεί που δεν εφαρμόζονται. Και να πω Βέλγιο, Αυστρία, Βέλγιο, Ελλάδα. Αυτέ είναι οι τρει χώρε που δεν έχουν ακόμη υπογράψει την συμφωνία. Σα παρακαλώ να το πράξουν τάχιστα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα έχει το λόγο η Επιτροπός. Ε, Κύριε Μάλστρον, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ευχόμενοι σε όλους ε, ευτυχισμένο τον καινούριο χρόνο και προσβλέπω σε στενή συνεργασία μαζί σας τους υπόλοιπους μήνες ε, στην Ολομέλεια και σε άλλε περιστάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή ΙΝΤΕ και του δύο συνεισηγητέ, τον κύριο Μπέκε και τον Σαντιάγο Φίσα, ε, για τις εκθέσεις ε, που μόλις ε, παρουσίασαν όσον αφορά την εφαρμογή του πυλώνα εμπορίου για τη Συμφωνία Σύνδεση με την Κεντρική Αμερική και τη Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ενώσεω και Περού και Κολομβία. Και οι δύο εκθέσει δίνουν πολύ σημαντική συνεισφορά για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των συμφωνιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση ξεκινά αυτό το χρόνο μια πλήρη αξιολόγηση και σχετική μελέτη για τι δύο συμφωνίε. Όπως σωστά είπατε στις εκθέσεις, η εφαρμογή πήγε καλά, η υλοποίηση πήγε καλά, είχε θετικό αντίκτυπο όσον αφορά το διμερές εμπόριο παρά τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει το δυσμενές διεθνές οικονομικό πλαίσιο. Θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα την υλοποίηση των διατάξεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε κάποιες χώρες Κεντρικής Αμερικής κυρίως όσον αφορά τις διατάξεις περί εργατικού δυναμικού και εργασίας. Όπως είπατε, επετεύχθη πρόοδος όσον αφορά τη δημιουργία του τριμερούς ε, Συμβουλίου Εργασία στην Γουατεμάλα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει χρήματα για εκδηλώσει για την εταιρική ευθύνη, για την ενίσχυση των εσωτερικών ομάδων παροχή συμβουλών και στα περιφερειακά γραφεία του Διεθνού Γραφείου Εργασία. Η Κολομβία και το Περού έκαναν κάποια πρόοδο όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων περιβιώσιμη ανάπτυξη. Η επαφή με το Περού ήταν ιδιαίτερα εντατική. Στον Υπουργό Εμπορίου ε, του Περού έστειλα επιστολή και ξέφρασα ανησυχία μου διότι δεν προστατευόταν επαρκώ τα εργασιακά δικαιώματα και τα, έχει χαλαρά, ε, χαλαρές προδιαγραφές το περιβάλλον για το εμπόριο και τις επενδύσεις στο Περού και δεν υπήρξε επαρκής διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών. Το Περού συζήτησε πολύ επικοδομητικά και έχουμε πετύχει θετικά αποτελέσματα. Η έκθεση όσον αφορά Τη συμφωνία τονίζει σωστά τη σημασία που έχει η διαβούλευση στην κοινωνία των πολιτών και εδώ έχουμε πετύχει πρόοδο. Πέρσι η Κολομβία δημιούργησε ειδική συμβουλευτική ομάδα και το Περού έχει δεσμευθεί να συζητήσει τα θέματα τα περιβαλλοντικά και τα εργασιακά στα πλαίσια των διαφόρων μηχανισμών διαβουλεύσεων στην κοινωνία των πολιτών που έχει επιλέξει η κυβέρνηση. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε ιδιαίτερα αυτό το τομέα και θα ερχόμαστε σε επαφή με αυτέ τι χώρε που καλύπτουν τι συμφωνίε σύμφωνα με το σχέδιο δράση με τα 15 σημεία για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη που παρουσιάστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Κάποια θέματα καλύπτονται μόνο εν μέρη σε αυτέ τι συμφωνίε ή δεν καλύπτονται καθόλου. Το θέμα του φύλου, ε, η καταπολέμηση του φυλου κατά καταπολεμηση διαφθορα και ένα κεφάλαιο για τι επενδύσει Βέβαια αυτό οφείλεται βασικά σε κάθε συμφωνία που σαν το 2010 και έληξαν διαπραγματεύσει τότε. Θα πρέπει να δούμε του εταίρου πώς μπορούμε να προχωρήσουμε όσον αφορά αυτά τα προβλήματα στο μέλλον. Τέλο, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι πλήρω συμφωνούμε με την άποψή σα. Πράγματι, υπό το φω τη προβληματική πολιτική καταστάσεω στην Κεντρική Αμερική και την περιοχή των Άνδεων, είναι κατεπίγουσα η ανάγκη και για θέμα αξιοπιστία, όπω είπατε κύριε Μπέγκε, σωστά, θα πρέπει και οι δύο συμφωνίε να τεθούν πλήρω σε ισχύ. Έτσι, υποστηρίζουμε ένθερμα το την έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε τα κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμα κυρώσει τη συμφωνία να το κάνουν το ταχύτερο δυνατόν. Προσβλέπω σε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Επίτροπε. Ο κύριος Αλαφράγκα έχει το λόγο για ένα λεπτό εν ονόματι του ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν συγχαρητήρια στους ε, εισηγητές για το έργο τους. Ε, ήμουν μάλιστα εισηγητής της Επιτροπής ΑΦΕΤ κατά την κύρωση των δύο συμφωνιών και χαίρομαι γιατί ήταν πολύ χρήσιμα εργαλεία για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών αυτών των άδειων και συνέβαλε σε, σε μία τάξη με κανόνες αποφεύγοντας προσταστευτικές τάσεις. Ε, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε λοιπόν τα πλεονεκτήματα των συμφωνιών και να βελτιώσουμε την εφαρμογή, όπως είπε ο κύριος ε, Μπέγκε. Είναι αδιανόητο ότι ακόμη τρεις χώρες μέλη δεν προέβησαν στην κύρωση αυτών των συμφωνιών, στην περίπτωση της Κολομβίας τα επιτεύγματα που επιτεύχθηκαν επισκιάστηκαν ε, από την ε, δινή κατάσταση της Βενεζουέλας. Πάντως χαιρετίζουμε την αποφασιστικότητα του Πρόεδρου που εξέφρασε την αλληλεγγύη του με τους δημοκράτες της Βενεζουέλας. Και επίσης ε, στα, στα θέματα της Κεντρικής Αμερικής μία αντιπροσωπή θα πάει στην Ικαράγουα για να διαπιστώσει αν η τραγική κατάσταση αυτή της χώρας συνάδει με τη δημοκρατική ρήτρα που συνήθως περιλαμβάνουν οι αντιστοιχείς εμπορικές συμφωνίες. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών, κυρία Ροντρίγκε Πινιέρο Φερνάνδε. Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ του δύο συγκητέ και να του τους ευχαριστήσω για την επικοδομητική του στάση, χάρη στην οποία καταλήξαμε σε ευρείε συμβαστικέ προτάσει. Σίγουρα πριν την εφαρμογή θα πρέπει να αξιολογήσουμε την προσωρινή εφαρμογή αυτών των συμφωνιών. Ε, οι συμφωνίε αυτέ έχουν κοινά σημεία με τι εμπορικέ μα συμφωνίε με τι υπόλοιπε χώρε τη Κεντρική Αμερική. Καταρχήν, έχει μια στρατηγική αξία. Ε, είναι υπέρ τη πολυμέρεια, τη παγκόσμια διακυβέρνηση και τη ε, περιφερειακή ολοκλήρωση, που είναι βασικοί πυλώνε τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η συμφωνία με την Κεντρική Αμερική είναι η πρώτη περιφερειακή συμφωνία που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι εμπορικέ συμφωνίε με το Περού και την Κολομβία, στι οποίε προσχώρησε και ο σημερινός ε, ακολουθεί ε, την ε, συμφωνία με τις χώρες των Άνδεων. Θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιηθούν οι νέες ευκαιρίες και να γίνει με μεγαλύτερη διαφοροποίηση αυτών των οικονομιών που είναι περιβολικά εξαρτημένες από τις πρώτες ύλες και τη γεωγραφική, γεωργική του συγγνώμη, παραγωγή. Θα ήθελα να τονίσω ότι και οι δύο συμφωνίες κατέληξαν σε μακροπρόθεσμες σε μακροπρόθεσμους συμβασμού και σε εμπορικούς κανόνες ε, που σέβονται πολύ περισσότερο τα εργασιακά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα. Επίσης, ε, η κοινωνία των πολιτών συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις ε, κάτι που θα ήταν αδιανόητο αν δεν υπήρχαν αυτές οι δύο εμπορικές συμφωνίες. Επίσης, χρειαζόταν χρειάστηκε η σύσταση ανεξάρτητων συμβουλευτικών ομάδων για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών στι συμφωνίε αυτέ. Γιατί όταν βλέπουμε ολόκληρα ανθρώπινα κύματα στην Κεντρική Ευρώπη να προσκρούν σε τύχη, όταν βλέπουμε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ικαράγουα ή όταν ζητούμε ρητή εφαρμογή τη Ενευτικής Συμφωνία της Κολομβίας, θα πρέπει να έχουμε επίγνωση πόσο σημαντικά είναι τα εφόδια που δίνουν οι εμπορικέ συμφωνίες και να φροντίσουμε να εφαρμοστούν πλήρω. Γι' αυτό, εκ μέρους των σοσιαλιστών, ζητώ τεράστιε προσπάθειε για να εφαρμοστούν πλήρω οι δύο συμφωνίε και να προσπαθήσουμε να τις καταστήσουμε πιο αποτελεσματικές, χωρίς αποκλεισμούς, με κεφάλαιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κεφάλαιο για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, ένα κεφάλαιο για το εμπόριο και το, την ισότητα των φύλων και επίσης να προβλέψουμε ένα μηχανισμό επιβολής κυρώσεων ως ε, ίστατο μέσο αν δεν ε, τηρηθεί η ρήτρα της βιώσιμης ανάπτυξης και μια επιπλέον ε, δέσμευση υπέρ της στήρησης συμφωνίας των Παρισίων. Εμείς ε, έχουμε κοινέ αξίε και αρχές με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και έχουμε πολλά να συμβάλλουμε προκειμένου να έχουμε ένα πιο δίκαιο εμπόριο και χωρίς αποκλεισμό. Ας βάλουμε τα δυνατά μας λοιπόν. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Η ε, Νάντια Χίρς τώρα έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η προώθηση μια εμπορική πολιτική που θα βασίζεται σε αξίε είναι μια από τι μεγαλύτερε επιτυχίε Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλο και περισσότερο βλέπουμε ε, μια φιλελεύθερη υπογραφή στην ανταγωνιστικότητα με την Ιαπωνία. Κλείσαμε την πιο ε, φιλόδοξη εμπορική συμφωνία και έχουμε διάφορα κεφάλαια όπως η βιωσιμότητα και οι δημόσιες προμήθειες ε, που ε, προωθούν μια σύγχρονη εμπορική πολιτική. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία με την Κολομβία και το Περού, έχει φτάσει ε, πλέον σε μια πολύ σημαντική φάση της εφαρμογής αυτής της συμφωνία. Θέλουμε να προωθήσουμε τα εργασιακά δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βλέπουμε να έχουμε πρόοδο σε αυτό το τομέα, αλλά και σε ό,τι αφορά τις ε, στρατηγικές αξίες της ε, Ευρώπης είναι σημαντικές στη Λατινική Αμερική όμως βλέπουμε επιθετική πίσδυση της Κίνας ε, που προσπαθεί να πάρει μερίδια αγοράς όμως δεν βασίζεται σε μια δίκαιη ούτε βασιζόμενη σε αρχές εμπορική πολιτική αυτή η στάση της Κίνας. Πρέπει λοιπόν να να προωθήσουμε εμείς ε, τις αξίες αυτές και μια σταθερή Κολομβία θα αποτελέσει ε, μια άγκυρα ασφάλεια για όλη την περιοχή. Τώρα ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να ξεχάσει ούτε τις άλλες περιοχές Λατινικής Αμερικής. Ό,τι αφορά τις εμπορικές σχέσεις δεν πηγαίνουν πάντα καλά τα πράγματα. Παραδείγματο χάρη δεν έχουν εξαντληθεί δεσμολικές ποσοστώσεις και υπάρχουν ευρωπαϊκά προϊόντα και υπηρεσίε που δεν έχουν πρόσβαση στις αγορές Κεντρικής Αμερικής. Θα πρέπει λοιπόν να να να βελτιώσουμε και περισσότερο τα πράγματα στο μέλλον. Ε, θέλουμε μια ισχυρότερες ε, εμπορικές σχέσεις. Είναι ένα σημαντικό λιθαράκι για να καταστήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορικό πρωταγωνιστή. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα έχει το λόγο για 1,5 λεπτό από την ομάδα των Πρασίνων η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε δεν είναι και τόσο ευχάριστο να συζητά κανείς ε, ε, τελείως διαφορετικές χώρες σε αυτή την κοινή συζήτηση. Κολομβία και Περού ε, αφενός, Κεντρική Αμερική αφετέρου και καλό θα ήταν να, διατηρήσουμε την παράδοση για ε, τις εκθέσεις ε, αυτές, δηλαδή να είναι απομονωμένη η συζήτηση ε, ώστε να μπορούμε να συζητάμε την κάθε χώρα σε βάθος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπέγκε για την πολύ ισορροπή αγαπημένη του έκθεση σε ό,τι αφορά την Κεντρική Αμερική. Βλέπουμε να περιλαμβάνει πολύ σημαντικές έννοιες, όπως για παράδειγμα την αναφορά στις ειδικέ ε, ζώνες παραγωγής ε, που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται και οι ενδείξεις. Τώρα, θα ήθελα να αναφέρω τη μεγάλη μου ανησυχία τη εξελίξη στη Γουατεμάλα. Ειδική Επιτροπή του ΟΗΕ κατά της ατιμορρησίας ε, ε, δεν, οι ε, αξιωματούχοι της απελάθηκαν. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ κακό για τη χώρα. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο αυστηροί με τέτοιου είδους εξέλιξη. Ό,τι αφορά τώρα την Κολομβία και το παιδιά την Κολομβία, καιρό είναι να ενεργοποιηθεί η ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν πάρα πολλέ δολοφονίε ακτιβιστών ανθρωπιστικών δικαιωμάτων. Θα ήθελα να μα πείτε τι γίνεται με τα συνδικάτα από το Περού, ε, τα οποία διαμαρτύρονται ε, σε ό,τι αφορά τον υποβασμό των περιβαλλοντικών ε, κοινωνικών προτύπων λόγω υποτίθεται ε, τη εμπορική συμφωνία. ποια είναι η συνέχεια που δίνει στο ενδιαφέρον αυτό, στην ενδιαφέρουσα αυτή καταγγελία από τα Περουβιανά Συνδικάτα Κομισιών. Ευχαριστώ. Συγγνώμη για τη διακοπή ο κύριος Σόλς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Το έτος 2019 ξεκίνησε εδώ και δύο εβδομάδες. Ήδη όμως έχουμε έξι δολοφονίες ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία. Είναι ένας αποτροπιαστικός απολογισμό του 2018, ο οποίο φαίνεται να συνεχίζεται. Ε, επομένως, πώς δεν περιλαμβάνει η Κομισιόν στον απολογισμό για τις εμπορικές σχέσεις με την Κολομβία και το Περού αυτά τα γεγονότα. Το κλίμα της βίας, της καταστολής ε, των δολοφονίων δολοφονιών δεν είναι κάτι δευτερεύον. Η εμπορική πολιτική μα βασίζεται σε αξίε. και αυτό χρειά απαιτεί σαφεί ε, ε, προσεγγίσεις και απαντήσει. Ε, πρέπει να ανασταλεί η εφαρμογή τη συμφωνία, εάν μέχρι να αποκατασταθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίση, μέχρι στιγμή δεν έχει φέρει και τόσα πολλά για τον πληθυσμό τη Κολομβίας αυτή η συμφωνία. Επίση, αν δεν δράσουμε, παραμένει δρανή η βία και η κατάλληλη μεγάλη των δικαιωμάτων ε, και η καταστροφή του περιβάλλοντο θα συνεχίσει. Και αυτό όχι μόνο στην Κολομβία, στι Άντε και την Κεντρική Αμερική. Και βλέπουμε τι έγινε με τον νέο πρόεδρο τη Βραζιλία, τον Μπολσονάρο. Έχουμε λοιπόν ε, ανησυχίε με τι αποφάσει. Ε, απειλούνται τα τροπικά δάση, απειλείται σύγκρουση με του αυτόχθονε. Και όλα αυτά έχουν μια διεθνή διάσταση. Ε, όταν βλέπουμε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραβίαση, μάλλον καταστροφή του περιβάλλοντος, να μην θεωρείται ε, σημαντικό, αυτό μας ανησυχεί. Ε, και πραγματικά έχει έρθει πλέον η στιγμή η Ευρώπη να στείλει ένα πάρα πολύ σαφές σήμα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, παρακαλώ να τηρείτε τον χρόνο αγόρευσης. Αγαπητοί συνάδελφοι, ένα λεπτό τώρα ε, Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι συμπληρωματικό στατικό που προσθέτουμε στο εκρηκτικό αυτό κοκτέιλ που στέθεται στα άλλα με τη συμφωνία του Μερκοσούρ και θα έχει τρομερέ συνέπειε για τη γεωργία μα και την αλληλεία μα, για τι υπεράκτιε περιοχέ μα, κυρίω την μπανάνα, τη ζάχαρη και το ρούμι και για την υγεία των καταναλωτών εν γέννη. Η Κολομβία, ξέρετε όλοι, είναι, δεν σέβεται ούτε τους κανόνες περιγυνής, ούτε για το περιβάλλον, ούτε τα δικαιώματα του ανθρώπου, ούτε του παιδιού, ούτε τα δικαιώματα του εργαζομένου. Οι συνδικαλιστές δολοφονούνται, τα καρτέλ των ναρκωτικών ευημερούν και ακόμα και η πρόσβαση στην υγεία είναι πάρα πολύ άνηση. Στο Περού περίπου 3 εκατομμύρια παιδιά από 6 μέχρι 17 εργάζονται έξω από κάθε νομικό πλαίσιο και χωρίς την παραμικρή κοινωνική προστασία αναπτύσσεται τελικά τη δουλεία, την πείνα σε αυτές τις τρίτες χώρες, καταστρέφεται την υγεία των συμπολιτών μας και καταστρέφεται όλη τον τομέα. Λοιπόν, τα απολώμα όλα. Δεν κάνετε τίποτα τελικά. Αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι υποφελήσεις και είναι κατά των λαών τελικά. Ευχαριστώ. Κυρία Αντρικένα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι. Το Περού είναι από τι χώρε της περιοχή που αναπτύσσουν τον ταχύτερο ε, ε, ρυθμό. Και η Κολομβία είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία τη Λατινική Αμερική. Γι' αυτό η εφαρμογή τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτέ τι χώρε είναι θεμελιώδη σημασία. Ε, υποστηρίζουμε ένθερμα τη Συμφωνία Ερήνευση για την Κολομβία και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει η εμπορική συμφωνία να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για να διευκολύνει την εφαρμογή τη Ειρηνευτική Συμφωνία. Και δύο χώρε έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ από την ανθρωπιστική κρίση στην Βενεζουέλα και οι δύο έχουν υποδεχτεί μεγάλο αριθμό μεταναστών και θα πρέπει αυτό να το εκτιμήσουμε. Από την άλλη πλευρά, η προσχώρηση του Εκουαδόρ σε αυτή τη συμφωνία, θετικό βήμα, ενώ η συμφωνία παραμένει ανοιχτή και στι άλλε χώρε τη περιοχή. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου, τον Σαντιάκο Φίσα, για την πλήρη αυτή έκθεση που καλύπτει το μίσο που πρέπει να δούμε μεγαλύτερη πρόοδο. Πέραν αυτού, δίνει πλήρη αναφορά των περιοχών που πρέπει να καλύπτονται όπω οι καταβολέ διαφθορά, η ξέπλυμα χρήματο και η φοροδιαφύγη. Πρέπει να καλύπτονται από τη συμφωνία. Όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν, να καλυφθούν από τη ρήτρα αναθεώρηση. Θα πρέπει λοιπόν να δράξουμε τι ευκαιρίε που μα παρουσιάζονται. Σα ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βάντερ έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Χωρί μικρόφωνο. Χωρί μικρόφωνο. Now. Αξιότιμη Επίτροπη, αξιότιμη Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εφαρμογή του, ε, συμφωνή, του Ρητράς Βιωσιμότητας ε, Κολομβίας Περού ε, δεν ε, λειτουργεί ε, ικανοποιητικά. Μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από το του 2019 ήδη έχουμε έξι θύματα ε, και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί τάχιστα. Μετά την υπογραφή αυτής της συμφωνίας, ε, καθήκον μας είναι να προωθήσουμε την εφαρμογή του κεφαλαίου της βιωσιμότητας, να την παρακολουθήσουμε την εφαρμογή δεν μπορούμε απλά ε, να είμαστε υπερήφανοι που έχουμε ένα ανωδικό χάρτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να έχουμε γράψει συμφωνίε σύνδεση και έπειτα να μην ε, ε, παρακολουθούμε την εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Άρα πρέπει να μιλάμε για την εφαρμογή και να λέμε και τα πράγματα με το όνομά του και να κατονομάζουμε τα προβλήματα χωρί κυρώσει, παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων δεν πρόκειται να υπάρξει επαρκή πρόοδο. Ε, χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει δυνατότητα επιβολή ε, κυρώσεων και στο κεφάλαιο για τη βιωσιμότητα. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ πολύ και τώρα. Σα ε, σας ευχαριστώ και που τρίσετε το, χρόνο σα Και τώρα η κυρία Σάντσεθ Καλντεντέι, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ενώ εμεί συζητούμε για το πώ θα χρησιμοποιήσουμε τι δεσμολογικέ προτιμήσει, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κεντρική Αμερική είναι τρομακτική, ανατριχιαστική. Ιδιαίτερα σοβαρέ είναι οι περιπτώσει τη Νικαράγουα, Γουατεμάλα και Ονδούρα. Ε, Κυρίω η απέλαση των μελών τη Διεθνού ε, Επιτροπή κατά τη Ατιμορρησία. Αυτό είναι πολύ δυσάρεστο για τη Γουατεμάλα και κάτι τέτοιο ωφελεί τι ε, οργανώσεις που επωφελούνται από τη διαφθορά και την ατιμορρησία. Και κρίμα που μερικές, ε, ε, από τους επωφελούμενους από την κατάσταση αυτή είναι πολυεθνικέ εταιρείε ή θηγατρικέ τους. Μάλιστα, οι τέτοιε συμφωνίε δείχνουν ε, το πρότυπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, το νεοφιλελεύθερο που θέτει το εμπόριο ε, στο κέντρο και όχι του ανθρώπους. Θα πρέπει επιτέλου να έχουμε δεσμευτικέ ρήτες για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Χαιρόμαστε που είναι σαφή η, διάταξη, η συμφωνία, αλλά δυστυχώς αποσιωπούμε την κατάσταση στην Κεντρική Αμερική σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα στη γη και τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών. Ευχαριστώ, κύριο Κολομπιέ, για ένα λεπτό. Για μια ακόμη φορά έχουμε την Ιωστή Εμπορική Συμφωνία, κυρία Πρόεδρε, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιας ε, περιφέρειας ε, ε, με τρίτες χώρες. Έχουμε τεράστιο εμπορικό έλλειμμα εις βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπορικές μας σχέσεις και εμπορικές ροές που επίσης είναι ελληματικές, χωρίς προστασία και με σφετερισμό των γεωγραφικών ενδείξεων των ε, ευρωπαϊκών προϊόντων. Ε, μπορεί να μην είναι ε, τόσο ασαφή όσο η συμφωνία του Μερκοσούρ, αλλά και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχουμε ξεκάθαρε διατάξει, γιατί και στη συμφωνία αυτή περιλαμβάνονται οι γενε, γενετικώς τροποποιημένοι του Μονσάντο και προϊόντα κρέατος που περνάνε από τον Ικαράγουα και επίσης έχουν γενετική τροποποίηση και που περνούν και από τη διόρυγα του Παναμά. Θα πρέπει επιτέλους να πούμε όχι σε μια τέτοια συμφωνία χάρη της, οικονο... της γεωργίας μας, της επιστηστικής ασφάλειας και της ανεξαρτησίας μας, καθώς και χάρη της προάσπισης των εμπορικών μας συμφερόντων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριος Μάτο, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτέ οι συμφωνίε είναι αξιέπαινε εφόσον προωθούν την περιφερειακή ολοκλήρωση μεταξύ κεντροαμερικανικών χωρών, όταν προωθούν ένα δίκαιο εμπόριο για όλου, όταν προωθούν τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Ο Σαντιάγο Φίσας είπε πολύ σωστά ότι ναι μεν ήταν επωφελής ε, η ε, συμφωνία για όλου. Όμω, ε, υπάρχουν εμβληματικά προϊόντα όπω η μπανάνα, η ζάχαρη κτλ. που πλήττονται στην περίπτωση τη Μπανάνα, ναι, μεν υπάρχουν ε, σε αντάλλαγμα κάποιε ρήτρε διασφάλισης και ένα μηχανισμό σταθεροποίηση ε, που ολοκληρώνεται φέτο και πρέπει να παραταθεί η ισχύ του, όμω μέχρι τώρα δεν ενεργοποιήθηκαν ποτέ αυτά, παρότι υπήρξαν ε, σημαντικέ υπερβάσει στα όρια. Το Σεπτέμβριο του 2018, Γουατεμόλα Νικάρο πέρασαν 3,49 και 102% και το Περού επίσης τα τελευταία τέσσερα χρόνια πέρασε, υπερεύει και αυτό ε, τα ανώτατα όρια. Αυτό όμως δεν, είχε, ε, δεν, δεν λήφθησαν υπόψη οι αρνητικές επιπτώσεις για τους Ευρωπαίους Μπανοπαραγούς και ελπίζω επομένως να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προς αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Από τους σοσιαλιστές ο κύριος ε, Χαουρέγη για... Ατόντο. Ευχαριστώ. Η Λατινική Αμερική είναι σημαντικό εταίρο Ευρωπαϊκή Ένωση, γεωπολιτικό εταίρο αλλά και εμπορικό εταίρο. Οι συμφωνίε αυτέ διευκολύνουν τι αμοιβέ μα σχέσει και ευχαριστώ του ε, δύο εισηγητέ που είχαν την ευφυα να μα προτείνουν ε, ένα προβληματισμό για τι ε, δύο εμπορικέ συμφωνίε. Εγώ θα μιλήσω για τη συμφωνία με την Κολομβία. Θα πρέπει να συνδεθεί άμεσα με την Ειρηνευτική Συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πιέσει την Κολομβιανή κυβέρνηση ώστε να αντιμετωπίσει αυτό το κύμα βίας εις βάρος ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάτι τέτοιο είναι ασύμβατο με μια οικονομική και πολιτική συμφωνία όπως αυτή που έχουμε με την Κολομβία. Θα πρέπει λοιπόν να συνδυάσουμε τις δύο συμφωνίες και πιστεύω ότι και για την Κεντρική Αμερική και ειδικά για την Ικαράγουα, την ε, Γουατεμάλα και την Οδούρα. Ε, πρόκειται για τρει πολύ φτωχέ χώρε με πολλά εσωτερικά προβλήματα. Θα πρέπει να βοηθήσουμε λοιπόν αυτέ τι τρει χώρε. Αντί να επιβάλλουμε κυρώσει, καλύτερα να τίνουμε χείρα βοηθεία. Οι χώρε αυτέ ε, χρειάζονται τι συμφωνίε ω μέσο για να εκδημοκρατιστούν πλήρω. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ο κύριος Βαβέντσα έχει το λόγο για ένα λεπτό για το ΕΛΚ η Λατινική Αμερική και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πολύ μεγάλο δυναμικό συνεργασία σε ένα φάσμα παγκοσμίων προβλημάτων και όσον αφορά το εμπόριο. Και θα πρέπει να ενισχύσουμε γι' αυτό τι σχέσει μα μέσω εκτεταμένου διαλόγου πολιτική, κοινωνική ένταξη, οικονομικών και εμπορικών σχέσεων. Όπω το βλέπουμε, το εμπόριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την περιοχή διπλασιάστηκε την τελευταία δεκαετία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προτιμησιακέ συμφωνίε με 26 από τι 33 χώρε από την κοινότητα της Λατινικής Αμερικής και των χωρών Καραϊβικής και τη Συμφωνία Ελευθέρου μπορείου με την Κολομβία και το Περού. Αυτές οι συμφωνίες προβλέπουν σταδιακή και κοινή απελευθέρωση μέσω πλήρους, δημιουργίας ενός χώρου πλήρους για, ελεύθερο εμπόριο. Οι στρατηγικές συμφων... αξίες της συμφωνίας ξεπερνούν το εμπόριο διότι προβλέπεται να δημιουργηθεί βάση για βαθύτερε σχέσει με οκροπρόθεσμη δέσμευση για ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνικά δικαιώματα, τα δικαιώματα των ηθαγενών λαών για του γεωργού και για το περιβάλλον προφανώ. Αυτό το εμπόριο, το αυξανόμενο, προσελκύει επενδύσεις σε αυτές τις χώρες και συνεπώς βοηθά τις τοπικές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να ενισχυθούν στην περιφερειακή τους αγορά και να μπορούν να ανταγωνιστούν διεθνώς. Επίσης αποτελεί ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, μπορέσει να αναπτυχθεί περισσότερο και να αποκομίσει περισσότερα γεωπολιτικά ε, ωφέλη. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος, ο κύριος Βάντεν Καντελάρ έχει το λόγο ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, σαν μέλος της Επιτροπής Γεωργίας, σαν ένα Βέλγος, χαίρομαι που έχω τη δυνατότητα να μιλήσω σε αυτή τη συζήτηση. Συμφωνούμε όσον αφορά το ελεύθερο εμπόριο και θέλουμε να αναπτύξουμε το εμπόριο με τους Λατινοαμερικανούς εταίρους μας. Αυτό το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά περιμένουμε τις ίδιες φιλοδοξίες από πλευρά των εταίρων μας. Και είναι τεράστια έκπληξη που διαπιστώνουμε ότι η Κολομβία δεν έχει σεβαστεί κάποιους ε, κανόνες, παραδείγματος χάρη, όσον αφορά ε, παγωμένα τηγανιτά προϊόντα. Ε, οι δασμοί είναι πάρα πολύ χαμηλοί, αλλά θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία όσον αφορά τις τηγανιτές πατάτες κατεψυγμένες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι καταστροφικό για τους εργαζομένους μας και τους πολίτες μας, διότι θα πρέπει να κάνουμε κάποιες προσαρμογές η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταστήσει σαφές ότι βοηθούμε όλες τις χώρες, μεγάλες και μικρές. Ε, αν δει κανεί ότι ένα γεωργό αντιμετωπίζεται άδικα, από εμά εξαρτάται να προστατεύσουμε αυτού του γεωργού που αδικούνται. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό θα πρέπει να το καταστήσει σαφές και θα πρέπει κατεπηγόντω να αντιμετωπιστούν όλα τα θέματα αυτό στο διεθνέ προσκήνιο. Σα ευχαριστούμε πολύ και τώρα περνάμε στη διαδικασία προσέλκυση προσοχή ε, του Προέδρου, Catch the Eye δηλαδή. Δεν έχουμε όμως και πάρα πολύ χρόνο. Έξι συνάδελφοι έχουν ε, ζητήσει να μιλήσουν. Ε, θα έχουν όλη τη δυνατότητα να το πράξουν. μιλά μόνο πρώτος. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Είναι... Ανέκαθεν ήμουν υπέρ της σημασίας, επεσήμανα τη σημασία που έχουν οι σχέσεις μας με τη Λατινική Αμερική. Είναι φυσική μας εταίροι χώρες αυτές. Γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας στο ισχύον πλαίσιο που υπάρχει μια έξαρση των προστατευτικών δυνάμεων, θα πρέπει να υπερασπίσουμε το πλεονέκτημα ισορροπημένων εμπορικών συναλλαγών που θα είναι αμοιβαίω υποφελή. Οι συμφωνίε με τι χώρε τη Λατινική Αμερική συμβάλλουν στην οικονομική του ανάπτυξη, στον εξυγχρονισμό των οικονομιών του και ταυτόχρονα στη διαφοροποίηση των εξαγωγών του σε ό,τι αφορά τι ευρωπαϊκέ χώρε. Και εμεί θα, ε, θα πρέπει να εξάγουμε τα προϊόντα μα. Δεν αυξάνεται ο πληθυσμό μα, αλλά ούτε και η εσωτερική κατανάλωση. Και λόγω τη κρίση, αλλά λόγω και τη αύξηση των δημοσίων δαπανών, λόγω τη ανάγκη ε, εξηγήσεων των οικονομικών. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε εξωτερικέ αγορέ για τι επιχειρήσει και την απασχόλησή μα. Επίση, θα ήθελα να ζητήσω για μία ακόμα φορά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την εμπορική συμφωνία με το Μερκοσούρ. Ε, η ε, Επίτροπο γνωρίζει πόσο ιστορική είναι η ευκαιρία που μας δίνεται και θα ήταν κρίμα να τη χάσουμε. Ευχαριστώ Λόπες Αγγελάρ για τους σοσιαλιστές για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Μάνστρομ, ως Ευρωπαίος Σοσιαλιστής είμαι ένθερμος υπέρμαχος ε, της Συμφωνίας Σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική με ρήτρα βιώσιμης ανάπτυξης, καταπολέμηση διαφθοράς ε, και ισότητα των φύλων. Και ω Ισπανό Σοσιαλιστό, επιφύλακτα ε, θέλω να έχουμε ω στρατηγικό εταίρο τη Λατινική Αμερική. Αλλά ω Σοσιαλιστή από τα Κανάρια, από αξόχω απόκεντρη περιοχή, θα ήθελα να εκφράσω την ανησυχία μου για τον αντίκτυπο που θα έχει σε ευαίσθητου τομεί αυτή η συμφωνία γιατί συνδυάζεται αυτή η συμφωνία με τον κανονισμό για τις ρήτρες διασφάλισης ε, που προβλέπει αντισταθμιστικά ωφέλη όταν έχουμε αρνητικό αντίκτυπο για τα ευαίσθητα προϊόντα των εξόχως απόκεντρων περιοχών γιατί τίποτα δεν βλάπτει ε, την εσωτερική ένωση όσο το διαζύγιο που προωθούμε και κάνουμε. Γιατί αν προσθέτουμε υποσχόμαστε αντισταθμίσει για ευαίσθητε περιοχέ που πλήττονται από εμπορικέ συμφωνίε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την υποχρέωση να προσφέρει αυτέ τι αντισταθμίσει και να μην αθέτει τι υποσχέσει τη. Σα ευχαριστώ, συνάδελφο κύριο Μαριά, για το ECR για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Συζητούμε τι ε, εμπορικέ συμφωνίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τι χώρε τη Λατινική Αμερική ε, και συμφωνίε σύνδεση αλλά είναι δεδομένο ότι πρέπει οι χώρες αυτές να τηρούν ορισμένα πρότυπα ορισμένες ρήτρες πρώτα απ' όλα την προστασία του περιβάλλοντος δεύτερον να διασφαλίζουν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επίσης τα εργασιακά στάνταρτς, διότι διαφορετικά έχουμε ένα έντονο κοινωνικό ντάμπινγκ. αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Ε, πρέπει επίσης να επιμείνει η ευρωπαϊκή ένωση να υπάρξει προστασία των ε, ντόπιων πληθυσμών να μην τους αρπάζουν τη γη να υπάρχει περιορισμός στην ασυδοσία των πολυεθνικών επιχειρήσεων και φυσικά να περάσουμε ένα μήνυμα ε, για την προστασία και την ισότητα των δύο φύλων. είναι προφανές ότι από τις τοποθετήσεις που υπήρξαν ότι υπάρχουν και αρνητικές επιπτώσεις και στην ευρωπαϊκή οικονομία. όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν οι συγκεκριμένες εμπορικές συμφωνίες. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα το λόγο έχει η κυρία Άννα Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. σε μια έκθεση με τέτοια χαρακτηριστικά και σε μια τέτοια συζήτηση για αυτέ τι περιοχέ του κόσμου, νομίζω ότι σοβαρό θα ήταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γίνει μια συζήτηση ξεχωριστά για την κάθε περιοχή, ε, για την κάθε εδαφική περιοχή και όχι μια κοινή συζήτηση. που δεν μπορεί να είναι τόσο ευρεία όσο θα άξιζε ε, για εμάς και για τους κατοίκους αυτών των χωρών ούτε και τόσο σοβαρό στην ομάδα μας. Μας φαίνεται το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε μια παρακολούθηση των εμπορικών συμφωνιών εφόσον αυτές έχουν ήδη συναυθεί ε, και λήξει ουσιαστικά. Εμείς θα θέλαμε αυτό να γίνεται στο πλαίσιο της εφαρμογής. Το 2013 ε, είχαμε αντίθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από μεγάλο μέρος ε, της ε, κοινωνίας των πολιτών σε κάποιες ρήτρες της συμφωνίας το 2013 και στον Παναμά δεν ε, παρουσιάζονται σωστά τα πράγματα ε, στην έκθεση. Παραδείγματο χάρη ε, δεν αναφέρεται το θέμα ότι είναι φορολογικό παράδεισο τα Panama Papers. Θα θέλαμε λοιπόν να αναθεωρηθεί. Επίση, καταπολέμηση τη διαφθορά, ξέπλυμα χρήματο, φοροαποφυγή. Πρέπει να αναφέρονται. τώρα, οι μπανάνες από την Ονδούρα ή ο κολομβιανός καφές μας αρέσει να τα απολαμβάνουν αυτά τα προϊόντα, αλλά κλείνουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας μπροστά στη φοροαποφυγή. Ευχαριστώ πολύ. Γκίγκολ, μάλλον Τζούλι Γόρντι τελευταία. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται συζήτηση για εμπορικέ ε, συμφωνίε χωρί να συζητούμε την πολύ ανησυχητική κατάσταση που επικρατεί στην Ικαράγουα όπου επιθέσεις κατά του ανεξάρτητου τύπου και των ε, επικριτικών φωνών της κοινωνίας των πολιτών είναι όλο και πιο έντονες, με απειλή απιλές και γνήσια βία κατά των δημοσιογράφων. Η ελευθερία του τύπου είναι από τους ακρογωνιαίους λήθους των δημοκρατιών και πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσει την πολιτική της επιρροή για να επιβάλλει την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα ανθρώπινα δικαιώματα στους εταίρους της. Πρέπει λοιπόν η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αξιοποιηθεί για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γιατί είναι το κατάλληλο μέσο γι' αυτό. Ωστόσο δεν βλέπουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει προτεραιότητες σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα στους επενδυτές ε, που προέρχονται από τους κόλπους της για να ζητήσει την, και πρέπει να ζητήσουμε κατεπηγόντως την ε, τήρηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Εμείς στο Κοινοβούλιο έχουμε υπερψηφίσει την θέση αυτή τον Οκτώβριο και γι' αυτό πρέπει να τηρήσουμε αυτά τα οποία εμείς οι ίδιοι έχουμε ζητήσει. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να καλωσορίσω όλους τους συναδέλφους που έφτασαν τώρα στην αίθουσα. Πριν ε, έρθω παρακολουθούσα στην τηλεόραση την ψηφοφορία στο Βρετανικό Κοινοβούλιο το οποίο απέρριψε τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου στο θέμα του Brexit. Επομένω θα συνεχιστούν οι συνομιλίες και ειδικότερα το ζήτημα της πρώτας μορφής κατά της κυβέρνησης ε, της Βρετανίας. Δεν ξέρω αν είχατε παρακολουθήσει τις εξελίξεις και γι' αυτό σας το αναφέρω. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Μάλστρομ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν συζητούμε σήμερα τη συμφωνία Μερκοσούρ. Γιατί δεν υπάρχει ακόμα τέτοια συμφωνία. Πολύ ευχαριστώ όμω όταν έρθει η ώρα και έχουμε ετοιμάσει τη συμφωνία, ε, θα έρθω να σα ε, την παρουσιάσω. Συζητούμε όμω αυτέ τι δύο συμφωνίε και το Κοινοβούλιο βέβαια έχει την αρμοδιότητα να οργανώνει τι ε, συζητήσει του σε μια περιφερειακή συμφωνία. Ίσως είναι δύσκολο να γίνει αναφορά σε κάθε χωριστή χώρα, αλλά πάλι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια διαδικασία για χωριστέ αξιολογήσει τη κάθε χώρας χωριστά. Άρα θα τις μελετήσουμε την καθεμία ξεχωριστά. Έχουν δώσει αποτελέσματα και σημαντικά αυτές ε, οι συμφωνίες. Πολλά όμως ακόμα μένουν να γίνουν και όπως είπαν και οι δύο εισηγητές πρέπει ιδιαίτερα να εστιαστούμε στην ε, υλοποίηση δουλειά. Πρέπει να γίνει ακόμη σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη προσοχή έχουμε δώσει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις χώρες που συζητούμε με ιδιαίτερη πληροφορία που τους απευθύνεται από τον ιστοτοπό μας, με τη βάση δεδομένων για την αγορά εργασίας, για, τα, για τους δασμούς, για τις στατιστικές, άλλες προϋποθέσεις που απαιτούνται. Και έτσι προσπαθούμε να φέρουμε σε επαφή τις ευρωπαϊκές με τις λατινοαμερικανικές επιχειρήσεις. Οι συμφωνίες αυτές είναι καλές κατά κάποιο τρόπο, όμως είναι και πεπαλαιωμένες. Ε, όντως ε, έχουν συναυθεί από το 2010, έχουν περάσει 10 χρόνια και τώρα πρέπει να προσθεθούν και άλλα καινούρια στοιχεία σε αυτές τις συμφωνίες. Έτσι λοιπόν μαζί με τους εταίρους μας θα ε, σκεφτούμε, θα μελετήσουμε πώς μπορούμε να εισαγάγουμε τα νέα αυτά στοιχεία σε μεταγενέστερο στάδιο. Υπάρχουν ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάποιες από τις χώρες αυτές. Συμφωνώ ότι είναι ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση στην Ικαράγουα, το έχουμε επισημάνει και πέραν αυτών των συμφωνιών βεβαίως υπάρχουν μέσα που, μπορούν, που μας επιτρέπουν να καλύψουμε και τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άλλωστε, οι Υπουργοί των Εξωτερικών την επόμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, έχουν συνεδρίαση όπου θα συζητήσουν και θα κάνουν και δήλωση για το θέμα αυτό ειδικά της Νικαράγουας. Στο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα επανέρχονται συνέχεια τα θέματα αυτά τακτικά στις επαφές μας με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ωστόσο δεν μπορούμε και να αρνηθούμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί με το Περού επί παραδείγματι, με το οποίο έχω συνομιλήσει συγκεκριμένα για το θέμα που επεσήμανε η κυρία Χάουταλα για τα εργασιακά ζητήματα, η οποία μάλιστα δεν είναι εδώ τώρα, ε, θέματα